σα διαβάσω μια μικρή παράγραφο που λέει ότι σε σχέση με την απόφαση πολλών επιτροπών προκειμένου να ξεκινήσουν ε, διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 69Γ, παράγραφος 1, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα 13 Μαρτίου, δεν ζητήθηκε ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, οι κοινοβουλευτικές αυτές επιτροπές μπορούν να μπουν στις διαπραγματεύσεις. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Υπάρχει διαδικαστικό από τον κύριο Κάρβερ όμως. Ένα λεπτό παρακαλώ για το διαδικαστικό σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις γύρισα από το Λονδίνο. Μετά από μια μικρή συνάντηση που είχαμε πρέσβει, ο οποίος εξηγεί την τραγωδία στην Αφρική, στην Κένια, όπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, πεθαίνουν από πείνα, και θα έπρεπε, μου ζήτησε να κάνω ό,τι μπορώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνειδητοποιήσουμε όλοι το τι συμβαίνει στο της Αφρικής και μου ζήτησε να φροντίσουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους εκεί. Ψηφοφορία. Έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα Σάντζεθ Νέιρε για τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αλλαγές ε, για την Κροατία μετά την προσχώρησή της. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία.